I Good morning, everybody. I think uh, we can start now. Mm, let me first. Η καλημερα Καλημέρα, καλώς ορίσατε πρώτα-πρώτα. Ε, ακόμα δεν έχει αρχίσει το, το εργαστήρι μας ε, Είμαι η Πάολα Φερνάντες, είμαι από την Ισπανία και θα σας τα πω όμως στα αγγλικά. Πάντως έχουμε διερμηνία έχουν αρχίσει να δουλεύουν οι διερμηνείς προς μια σειρά γλωσσών, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, εστονικά, ιταλικά, ε, ολλανδικά, σλοβακικά, σουηδικά και προς ελληνικά, αλλά δεν το αναφέρει πρόεδρος. Οπότε μπορεί να ακούσετε σε αυτές τις γλώσσες τη μετάφραση. Και τώρα να πούμε τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την σημερινή ημέρα. Έχουμε σε αυτό το προσαγωγικό τμήμα, ένα τεταρτάκι και η επίσημη έναρξη της συνάντησης θα γίνει στις 11 η ώρα. Θα έρθει ο Γενικός Διευθυντής για την επικοινωνία αλλά και ο ε, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή Αντιπρόεδρος που είναι αρμόδια για τα θέματα ισότητα των φύλων και έτσι θα δούμε πώς θα συγκροτηθούν τα, τα πάνελ της, ε, για τη συζήτηση, θα έρθουν ευρωβουλευτές, ε, εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με τα σημερινά μας θέματα. Και επομένως, ο πλευράς πρακτικής. Να σας πω κάποιες λεπτομέρειες πριν δώσω τη σκητάλη στους στις συναδέλφους που είναι εδώ. Έχετε λάβει ένα ντοσχέ με το πρόγραμμα, το, το, υλικό γενικότερα, ό,τι θα χρειαστεί εδώ για να συζητήσουμε τα θέματα της Επιτροπής γυναικών, έχετε τα βιογραφικά των βουλευτών, διάφορες ιστορικές πληροφορίες. Επίσης έχετε λάβει υλικό πολύ από το email και από το Ευρωβαρόμετρο επίσης κάποιο υλικό το οποίο σήμερα θα συζητήσουμε. As the, very big news event of the day. Uh, in order to... Επίσης, για να μπορέσουμε να, στείλουμε την ενημέρωση με mail θα σας μοιράσουμε ένα φιλοχαρτίο που θα πρέπει εκεί να γράψετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και εκεί θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να λαμβάνετε και ενημέρωση για τις δραστηριότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε, εκεί ή θα τσεκάρετε στο κουτάκι με την πλασχετική ερώτηση ή όχι και εμείς αντιστοίχως θα σα ενημερώνουμε ή όχι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, τώρα ε, μας πιέζει ο χρόνος. Και θέλω να μου πείτε αν έχετε κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά αυτά τα πρακτικά ζητήματα. Ε, Επίσης, αν κάτι προκύψει, μπορεί να με βρείτε εδώ γύρω-γύρω. Έχουμε το Walter, έχουμε ένα σωρό άλλου υπαλλήλους από την υπηρεσία μας εδώ του Κοινοβουλίου, ε, που οργανώσαμε αυτή τη συνάντηση και τώρα προχωρούμε. Και θα δώσω τον λόγο στις συναδέλφους. Βρισκόμαστε εδώ ε, και θα μείνουμε εδώ αλλά ίσως ε, δεν πειράζει τώρα αλλά όταν αρχίσει το κυρίως τμήμα της συνάντησης ίσως μπορείτε να έρθετε λίγο πιο κοντά να κάτσετε εδώ στα μπροστινά έδρανα, για να μπορώ να σας διακρίνω και εγώ καλύτερα. Καλά, ό,τι θέλετε κάντε τέλος πάντων. Τώρα. Ντουάτ είναι, είναι η συνάδελφος δεξιά μου που είναι η επικεφαλής η, ε, της, ε, η πρόεδρος της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων. Οπότε θα μας ενημερώσει σε σχέση με το τι δραστηριότητες έχουμε αναπτύξει τώρα τελευταία, Σαμπίνα Μανιάνο επίσης, από την Επιτροπή και θα σας εξηγήσει και αυτή κάποια τέτοια σχετικά ζητήματα, να σας πει ποια νομοθετήματα έχουν επεξεργαστεί στην Επιτροπή αυτή. Ε, φυσικά θέματα που έχουν σχέση με την ισότητα των ευκαιριών. Έχεις το λόγο. Με δύο λόγια, μια που πιέζει ο χρόνος, να σας τα πω. Η Επιτροπή των δικαιωμάτων της γυναίκας ασχολείται με θέματα ισότητας των φίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής. Έχει αυτή την εντολή. Επίσης, έχει αναλάβει την, την, το mainstream, δηλαδή την ένταξη των θεμάτων των γυναικείων στις υπόλοιπες πολιτικές ένωσες. Ε, θα έρθει και η κυρία Μπάουρα να σας τα πει, που είναι, έχει αναλάβει κάποια σημαντικά ζητήματα και επομένως ε, θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει νομοθεσία για τα θέματά μας. Ε, έχουμε και άλλα βέβαια που μας απασχολούν. Να, φέτος ε, θα ασχοληθούμε με τις εργασιακές συνθήκες ε, των γυναικών στον κλάδο παροχή υπηρεσιών, για την σχέση με την πράσινη οικονομία, τι γίνεται στι τρίτε χώρε, τι γίνεται στην Βόρεια Αφρική, τι γίνεται στα Βαλκάνια, στι χώρε που βρίσκονται σε πρωταξιακό καθεστώ και επομένω βλέπετε πόσο ευρία είναι η εντολή τη Επιτροπή μα τώρα. Σε σχέση με τι άλλε επιτροπέ, έχουμε ότι για θέματα νομοθεσία όσον αφορά την προστασία των γυναικών θυμάτων. Άρα συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών και, ε, και άλλες, ε, οπότε προσπαθούμε να δούμε πώς θα προστατευτούν τα θύματα της ε, οικογενειακής οικιακής βίας, οπότε συνεργαζόμαστε και με την Επιτροπή Απασχόλησης, ούτως ώστε να θεσπίζεται αρτιότερη νομοθεσία για τις ε, γυναίκες στα εργασιακά. Τώρα, δεν θα υπησιάδω σε λεπτομέρειες, δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση. Ε, από πλευρά τη επικοινωνία τώρα ξέρω ότι έχουμε ένα website το οποίο ενημερώνεται πάρα πολύ καλά. Έχουμε και ένα newsletter, είμαστε και στο facebook. Ευχαριστώ να απαντήσουμε οτιδήποτε ερώτηση. Σαβίνα, you want to add on this? Yes, maybe just a few words uh, on the connection η Σαμπίνα. Να σα πω τώρα για τη σχέση ε, των δύο αυτών επιτροπών. Αυτή που ασχολείται με την πολιτική απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα. Κοινωνική πολιτική, επομένω, ε, ε, αυτέ είναι οι βασικέ αρμοδιότητε και η Επιτροπή Επομένω Απασχόληση επίση ασχολείται και με τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη δυσμενή διακρίση, το χώρο εργασία, την αγορά εργασία γενικότερα και ακριβώ εδώ πέρα είναι ο κοινό τόπο σε σχέση με την Επιτροπή των Γυναικών ε, όπως σας εξήγησε η συνάδελφος, είναι μια από τις της ε, Επιτροπής μας. Ε, αυτού του είδους η, η... το να υπάρχει ισότητα για ίση δουλειά, ίση αμοιβή. Οπότε συνεχόμαστε πάρα πολύ στενά, ε, επεξεργαζόμαστε διάφορες ε, γνωμοδοτήσεις, και θα δείτε στο δεύτερο και στο τρίτο πάνελ συζήτηση θα συζητηθεί το τι γίνεται με την ε, νομοθεσία και μπορεί να δείτε εκεί ότι ε, θα υπάρχουν ε, βουλευτές και από τις δύο επιτροπές και η κυρία Ζήμερ που έχει αναλάβει μια έκθεση σχετικά με αυτό το θέμα. Τώρα, το θέμα το πώς θα γεφυρωθεί το μισθολογικό χάσμα, τι θα γίνει επίσης και με τις συντάξεις. Σίγουρα και η ανισότητα ε, που ισχύει στα μισθολογικά ισχύει και για τις συντάξεις. Είναι μοίρια συνέπεια και αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Απασχόλησης. Εμείς ασχολούμαστε με αυτά εδώ και πολύ καιρό και τώρα προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει με την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας όσον αφορά το έγγραφο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για η κυρία Ομινρόιτεν που είναι η, η συγγήτρια θα εμφανιστεί στο δεύτερο πάνελ να σας τα πει και τελικά θα καταλήξουν σε μια γνωμοδότηση. Επίσης, έχουμε την κυρία Ματέρα, που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Δικαιωμάτων των Γυναικών. Εκείνη, επίσης, είχε αναλάβει ε, μια άλλη έκθεση και αυτή θα πάει στο δεύτερο πάνελ. Βεβαίως, οι ανισότητε που διώκουν τη σχέση των δύο φύλων και στη συγκεκριμένη στην αγορά εργασία είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ε, πολιτική αυτή ισότητα. Ακόμα μας περιμένει πολλή δουλειά μπροστά μας. Πολλά επιμέρου ζητήματα γεννώνται και υπάρχει η κατανομή εργασία, αλλά τέλο πάντων να σα πω ότι η στόχη μα είναι κοινή. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, να σα πω τι έχετε λάβει σε αυτό το ντοσιέ. Έχετε λάβει το ψήφισμα μεταξύ άλλων που αφορά την έκθεση της Σοφία Ινετφέλτ. Πρόκειται για ένα ψήφισμα το οποίο την τελευταία εβδομάδα εγκρίθηκε στην Επιτροπή μα και πρόκειται να υποβληθεί στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Πρόκειται για ένα ψήφισμα πολιτικού χαρακτήρα. Εδώ θίγονται ένα σωρό ζητήματα τα οποία και θα συζητήσουμε σήμερα. και λοιπόν. Έχουμε και κάποια άλλη έκθεση ε, που σα ανέφερε η Αμέλ. Είναι κάποια ειδική διαδικασία που τη διέπει. Είναι το σχέδιο έκθεσης για την ίση αμοιβή. Αυτό λέει που συζητάμε σήμερα. Είναι η έκθεση Bauer. Η έκθεση Bauer ακόμα δεν έχει εγκριθεί στην Επιτροπή. Πρόκειται για τις προτάσεις της ε, συγκεντρίας. Σήμερα επομένω. όσα συζητήσουμε και αυτό θα αποτελέσει συμβολή στην έκθεση. Νομοθετική πρωτοβουλία δύο λεπτά και μας μένει, οπότε Αλμέλ, πες μας δύο λόγια γι' αυτό. Να σας πω. Πολύ σημαντική είναι αυτή η έκθεση για μας και για το περιεχόμενο, αλλά και πλευρά θεσμική. Όπως ενδεχομένω γνωρίζετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας και ε, υποβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση νομοθετική δεν είναι σαν ε, τα κράτη-μέλη όπου έχει κανεί την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο. Η συνθήκη προβλέπει ότι το δικαίωμα πρωτοβουλία το έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μπορούμε όμω εμεί στο κοινοβούλιο να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, κατεβάσει μια πρόταση. Και πριν από τρία χρόνια η προηγούμενη συνθήκη ε, έδινε λιγότερα δικαιώματα στο Κοινοβούλιο. Τώρα, επομένως, επομένως το Κοινοβούλιο μπορεί να, να ζητήσει ενώ πριν δεν μπορούσε να το ζητήσει εξίσου, τώρα να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαμορφώσει μια νομοθετική πρόταση. Και το ακριβώ το ίδιο έγινε τώρα και όσον αφορά την ισότητα αμοιβή. Δεν έχει ψηφιστεί, όπω είπαμε, το κείμενο αυτό στην ε, Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, διότι περιμένουμε να δούμε τι θα βγει, τι θα βγει σήμερα. Ο εισηγητή, η εισηγήτρια, οι σκιώδει εισηγητέ θα σα ε, συναντήσουν, θα τα πείτε, οπότε θα λάβουν υπόψη θα τους πείτε και έτσι επομένω, θα ολοκληρωθεί η δουλειά τους και θα παραπευθεί στην Αρμόδια Επιτροπή για έγκριση. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν ξέρω, έχουμε ώρα, έχουμε ερωτήσεις για πρακτικά θέματα. Αν δεν έχετε κάποια ερώτηση, τότε να δούμε εδώ να γίνει ε, το επόμενο πάνελ, να λάβουμε, να λάβουμε θέσεις. Και έχουμε επίσης και την Ευρένη συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό θα γίνει αύριο το πρωί. Και εκεί θα ζητηθούν τα σημερινά μας θέματα. Είναι ανοιχτή η κοινή συνεδρίαση και όποιος θέλει μπορεί να πάει. Τρία πάνελ. Και στο ημικύκλιο, εμπειρογνώμονες, εθνικοί βουλευτές, θα μας πούνε ε, ο καθένας από πλευράς που λέει τα πράγματα, αλλά θα έρθει και η Επίτροπος Ρέντιν και θα κλείσουμε με τον Τούρκο Υπουργό για τα Ευρωπαϊκά θέματα και το θέμα είναι ότι ακριβώς η Τουρκία ε, έχει πάρα πολύ μεγάλα, μεγάλο χάσμα διαφοράς μεταξύ των μισθών των ΜΕΝ και των ΔΕ. Πρώτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και τώρα προχωρούμε. Προχωρούμε τώρα στο επίσημο τμήμα της ε, συνάντησής μας. Τώρα θα δείτε ένα φιλμάκι. Βάζω και σας μην απολαύσετε την ταινία. Αυτό το φιλμάκι το έφτιαξε Γενική Διεύθυνση για την Επικοινωνία. Μπορείτε ελεύθερα να το απολαύσετε και στο ίντερνετ. Το link το έχετε λάβει στα έγγραφα του φακέλου. Όποιο θέλει μπορεί να το δει, να το χρησιμοποιήσει για δραστηριότητε ε, επικοινωνία. Τώρα αλλάζουμε θέση. Όποιο θέλει μπορεί να έρθει πιο κοντά. Τώρα, τώρα θα διαμορφώσουμε τη σύνδεση του επόμενου πάνελ. Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη μου ευχαρίστηση το να κηρύσω την έναρξη αυτού του σεμιναρίου. Είναι πάρα πολύ σημαντική η μέρα αυτή για όλους, όλες εμάς. Όλους και όλες λέω γιατί και άντρες και γυναίκες έχουμε ευθύνη ε, κοινή όσον αφορά το πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την υπόθεση της ισότητας. Χουάνα Σάντζεθ ονομάζομαι. Ε, ε έχω παντευτεί Βέλγο, ο οποίο ονομάζεται Λαού. Ε, και οπότε πάρα πολύ εδώ στο κοινοβούλιο με ξέρουν με το επίθετο του άντρα μου. Ε, δίπλα μου εδώ στα αριστερά μου είναι η Σιλβάνα Ε, πάρα πολλά χρόνια ήταν αντιπρόσωπο του κοινοβούλιο και επίση είχε αναλάβει τα θέματα τη ισότητα επί πολύ, πολύ καιρό. Και φυσικά ελπίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει μαζί τη ε, για μένα είναι κάπως αξιοπερίεργο ε, το να συζητούμε για ίση αμοιβή, για ίση δουλειά, γιατί αυτό διότι όλο ένα και περισσότερο αυτό το θέμα συζητείται και θα έπρεπε επομένω να μην υπάρχει πια πρόβλημα ε, μια που έχουμε τόση πρόοδο σημειώσει στα θέματα της ισότητας γενικά. Όμως, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Οπότε, τουλάχιστον για μας τις γυναίκες, παραμένει αυτό πηγή ανησυχίας όσον αφορά τον επαγγελματικό μας βίο. Και όπως μπορείτε να δείτε υπάρχει διερμηνία προς μια σειρά γλωσσών. Επομένως μπορείτε να μιλήσετε τη γλώσσα σας, μπορείτε να αποβάλλετε ερωτήσεις τη γλώσσα σας και επομένω, ε, όσο περισσότερο μιλήσουν, τόσο πιο ενδιαφέρουσα θα είναι η συμμετοχή, ζωντανή συνάντηση. Και βεβαίω, ελπίζω ότι θα γίνει σε, μέσα σε οικοδομητικό κλίμα η συνάντηση. Οι γυναίκε άλλωστε δεν δεκνόμαστε από θετικότητα. Σελβάνα, στα γαλλικά. Σήμερα το πρωί θα είναι εδώ και η Ρομπέρτα Αντζελίλη που είναι αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου και εκείνη και εκείνη επίση ασχολείται με τα θέματα ισότητα των δύο φίλων Όμω, δυστυχώ, για λόγου ανεξάρτητους από θέλησή δεν μπόρεσε να έρθει στην ώρα της, θα καθυστερήσει. και νομίζω ότι παρά το δεν έχει έρθει εδώ μπορούμε να αρχίσουμε. Έχεις το λόγο Σιλβάνα για να διευθύνεις αυτό το δεύτερο τμήμα του σεμινάριου. Herzlichen Dank, Juana, und herzlichen Dank für die Einführung. Herzlich willkommen alle hier. Ευχαριστώ πολύ για τα εισαγωγικά σχόλια. Ελπίζω να έχουμε χρήσιμες ε, συζητήσεις, ε, πλούσιες συζητήσεις. Η παράδοση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να έχουμε ανταλλαγές απόψεων με δημοσιογράφους ε, και με άλλα μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Για μας το θέμα της ίσης μεταχείρισης των ίσων ευκαιριών είναι ένα κεντρικό θέμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε και εγώ θα με αυτό το πρώτο εργαστήριο, το πρώτο πάνελ και θα σας αναφέρω κάποια σημεία τα οποία μας απασχόλησαν στην ε, ομάδα εργασίας που είχαμε με την ε, Ρομπέρτα Αντζελίλη. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητούμε εδώ και αρκετό ε, καιρό επεξεργαζόμαστε το θέμα της ίσης μεταχείρισης ε, και της ισότητας ε, των φύλων από πολλές απόψεις. Όποιοι και να είναι, αν θέλετε, η οπτική γωνία από την οποία κανείς ε, θέλει να εξετάσει το θέμα της ισότητας των φύλων και ανεξάρτητα από το αν το συζητάει κανείς στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή κάποιων άλλων, αν θέλετε, θεμάτων και τομέων, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι σε όλες τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας απασχολεί το θέμα της ισότητας, διότι βεβαίως πάντα υπάρχει κάποιος, ένα μέλος του Προεδρείου, ή ένα μέλος Επιτροπής που εγείρει το θέμα αυτό και το θέτει για τον ένα ή τον άλλο τομέα. Βεβαίως ε, συνεχίζουν να υπάρχουν κάποια θέματα που δεν έχουν ε, αρχικά τεθεί. Στη Γερμανία λέμε συχνά ότι αν κάποιος θέλει να αλλάξει τον κόσμο πρέπει να ξεκινήσει αλλάζοντας τον εαυτό του. Και βεβαίως θέλουμε να ξεκινήσουμε με κάποιες ε, αλλαγές εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παραδείγματος χάρη, πόσες γυναίκες βρίσκονται σε σημαντικές θέσεις, πόσες γυναίκες είναι επικεφαλής αντιπροσωπιών, επιτροπών, είτε στο Προεδρείο, μέλη του Προεδρείου, ε, αντιπρόεδροι. Και βεβαίως ε, προετοιμάζουμε κάθε φορά δραστηριότητες ε, οι οποίες θα ευαισθητοποιήσουν όλους όσους βρίσκονται ακόμα μακριά από αυτό το θέμα της, ε, των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων. Έχουμε εδώ και μία μπροσούρα, φαντάζομαι την έχετε όλοι στις, ε, στους φακέλους σας, με διάφορα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά την σύσταση των ε, διαφόρων επιτροπών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταρχήν και το Βέλγιο, λέει εδώ, Ε, δεν θυμάμαι τώρα ποιες άλλες χώρες, πέντε χώρες σε πάση περιπτώσει, όπου υπάρχουν πολλές γυναίκες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μάλιστα περισσότερες γυναίκες εδώ από ότι στις εθνικές βουλές. Μάλτα, Πολωνία, Βέλγιο. Θα δείτε τις υπόλοιπες χώρες αυτή την προσούρα και όπως ξέρετε από την πρώτη φορά που εξελέγει με άμεσες εκλογές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ποσοστό των γυναικών αυξήθηκε, 34% είμαστε, έχουμε φτάσει σήμερα και σε κάποιες περιπτώσεις 36% συμπεριλαμβάνουμε εδώ και βεβαίως και τις γυναίκες που βρίσκονται στο Προεδρείο των ε, επιτροπών. Η Οικονομική Επιτροπή, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή σημαντικής οικονομικής κρίσης. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν ε, τομείς ε, στους οποίους ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει η εκπροσώπηση των γυναικών και τα τελευταία χρόνια είδαμε σημαντικές μεταβολές στις γενικές διευθύνσεις. Τέσσερις γενικές διευθύντριες είναι γυναίκες σήμερα. Και αυτό είναι κάτι που έγινε τα τελευταία χρόνια. Γυναίκες λοιπόν συνεργάτες οι οποίες, ε, τον οποίων ο αριθμός διαρκώς αυξάνεται οι ενδιάμεσες ε, κατηγορίες διοικητικών θέσεων επίσης Συνεχίζουν ε, να υπάρχουν βεβαίως ε, διαφορές και στις ε, ανώτερες και στις μεσαίες κατηγορίες. Αν πάμε στις χαμηλές κατηγορίες, εκεί οι γυναίκες εκπροσωπούνται πιο σημαντικά. Αυτό που μας ενδιαφέρει βεβαίως είναι οι μεσαίες διοικητικές θέσεις, αυτές στις οποίες ακόμα οι γυναίκες δεν εκπροσωπούνται αρκετά. Βεβαίως υπάρχει το κεντρικό θέμα του πώς κανείς ε, μπορεί να συνδυάσει την οικογενειακή του ζωή με την επαγγελματική του ζωή. Αλλά αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σήμερα ότι δεν θα πρέπει να είναι μόνο μια απασχόληση, μια ανησυχία των γυναικών. Ε, υπάρχουν και άνδρες οι οποίοι όλο και περισσότερο αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Και δεν είναι μόνο οι γυναίκες σήμερα που προσπαθούν να συνδυάσουν, να συγκεράσουν την προσωπική του ζωή, την οικογενειακή του ζωή και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Και δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση ε, για κάποιον ο οποίος αντιμετωπίζει ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Το θέμα βεβαίως είναι και το θέμα των αποδοχών. Οι γυναίκες πολλές φορές έχουν διακεκομένες και διακεκομένες σταδιοδρομίες και πολλές φορές βλέπουμε ότι αναγκάζονται να σταματήσουν για κάποια σημαντικά χρονικά ε, διαστήματα την επαγγελματική τους δραστηριότητα για να ασχοληθούν περισσότερο με τις οικογένειες, με τα παιδιά τους. Το συνεχίζει να είναι κυρίως φαινόμενο που απασχολεί τις γυναίκες. Οι διακεκομένες αυτές τα διαδρομίες συνεχίζουν να είναι κυρίως ε, γυναικείες ε, καριέρες και στα σταδιοδρομίες. Ύστερα λοιπόν μπορούμε σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Η Χουάνα Λαρούς, η οποία είναι Γενική Διευθύντρια για θέματα επικοινωνίας, υπεύθυνη για τα θέματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. μπορούμε να συνεχίσουμε με την παρουσίασή της. Ευχαριστώ πολύ Σιλβάνα για την παρουσίαση που μας έκανες. Είναι πολύ χαρακτηριστική. Ευχαριστώ όλα τα μέλη που μας βοήθησαν σε όλη αυτή την εργασία. Σας καλωσορίζω όλους. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ισότητας των φύλων και της, των ίσων ευκαιριών. Άνδρες και γυναίκες θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες προαγωγής και εξέλιξης. Βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι κύκλοι βιολογικοί, φυσικοί, οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί να καθυστερήσουν τη σταδιοδρομία μιας γυναίκας. Ε, αλλά όχι μόνο, όπως παραδείγματο χάρη το πώς κανείς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα και ικανοποιητικά την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν οι μετακινήσεις, παραδείγματο χάρη, τακτικές μετακινήσεις στο Στρασβούργο. Κάτι που διαταράσει πολλές φορές την ζωή των γυναικών ή των γονέων που εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ερώτημα τι κάνουμε με τα παιδιά μας, τι κάνουμε την εβδομάδα αυτή το μήνα, δηλαδή 12 εβδομάδες το χρόνο που πρέπει να λείπουμε στο Στρασβούργο. Και πολλές φορές ε, πρόκειται για γονείς οι οποίοι ζουν στις Βρυξέλλες χωρίς να έχουν οικογενειακό και κοινωνικό ιστό. Οι περισσότεροι από εμά είναι ξεριζωμένοι, δεν έχουν τις οικογένειές τους και πολλές φορές ε, δεν έχουν ε, και τις δυνατότητες ε, να να αναθέσουν τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια αυτών των μετακινήσεων. Πολλές φορές δεν υπάρχουν και βρεφονιπιακοί σταθμοί ή αρκετές θέσεις. Καλωσορίζω όμως αυτή τη στιγμή την κυρία Κράτσα, η οποία ήταν αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου αρμόδια για θέματα επικοινωνίας. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η βοήθειά της, η στήριξή της και νομίζω ότι θα συνεισφέρει επικοδομητικά στην σημερινή μας συζήτηση. Έχετε το λόγο, όποιος θέλει να πάρει το λόγο. Βλέπω ότι κάποιος ζητάει το λόγο. Θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε μία σύντομη παρουσίαση. Ποιοι είστε πριν κάνετε την ερώτησή σας. Λέγομαι Ραφαέλ Πόρτο Καρέρο και να βρούμε στην ε, Φλαμαν... στο Φλαμανόφωνο τύπο στο Βέλγιο. Θα ήθελα να ξέρω πώς έχει η ισότητα των φύλων μεταξύ των διερμηνέων. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά σίγουρα, αν ε, κάνω λάθος, θα με διορθώσουν οι συνάδελφοι. Γνωρίζω τον τομέα αυτό αρκετά καλά. Δεν υπάρχει ούτε ευμενής ούτε δυσμενής ε, διάκριση. Όλοι όσοι εργάζονται εδώ περνάνε από τις ίδιες εξετάσεις και δεν υπάρχει καμία απολύτως, ε, αν θέλετε, βούληση στρατηγική να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες. Ε, εάν ε, στους διερμηνείς υπάρχουν περισσότερες γυναίκες και κοιτώ τις συναδέλφους στις καμπίνες των διερμηνέων, αυτό ίσως οφείλεται σε κάτι που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κάποια άλλη φορά, που είναι το θέμα της ε, πρόσβασης σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες σχολών, πανεπιστημίων και σπουδών. Γιατί υπάρχουν περισσότερες ή λιγότερες γυναίκες στα λεγόμενα ανδρικά επαγγέλματα ή σε κάποιες επαγγελ, ε, επαγγελματικές κατηγορίες ή σπουδές, επιστημονικές σπουδές. Οι συνάδελφοι διερμηνείς γνωρίζουν πολύ καλά ότι γνωρίζω το επάγγελμα της διερμηνίας. Πριν από πολλά χρόνια κάποια διευθύντρια η υπηρεσία διερμηνίας είχε πει, όχι εδώ στο Κοινοβούλιο, ότι όπως όλες οι γυναίκες ξέρουν να μαγειρεύουν, αλλά οι μεγάλοι μάγειροι και σεφ είναι άντρες, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την διερμηνία. Αυτό το θεωρώ πραγματικά διακριτικό και καθόλου ορθό. Η Ρομπέρτα Αντζελίλη όμως μόλις μπήκε στην αίθουσα, θα της παραχωρήσω αμέσως ε, τη θέση μου έτσι ώστε να μας παρουσιάσει το θέμα για το οποίο είναι σήμερα εδώ. Και βεβαίως πριν δώσω το λόγο στην κυρία Αντζελίλη, θα ήθελα να ρωτήσω τους διερμηνείς αν συμφωνούν με αυτό που είπα. Oui. Oui, bonjour, merci. Ε, Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα eh, Καλημέρα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, ε, την Γενική Διευθύντρια, του συναδέλφους, την κυρία Μένιν που ήταν η προκάτοχός μου διότι είμαι εγώ πλέον υπεύθυνη ε, στην ομάδα εργασίας για την ισότητα των δύο φύλων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια πράγματα. Όλοι έχουμε επίγνωση των διακρίσεων και της ανισότητας που επικρατεί ακόμη και σήμερα. Παρατηρείται μεγάλη ανισότητα σε διάφορες περιοχές του κόσμου και δυστυχώς θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα δικαιώματα των, ε, που αναγνωρίζονται στα δύο φύλλα, ε, ε, ιδίω δε σε κάποιους κλάδους. Η μεγαλύτερη διαφορά από όλες εντοπίζεται στην μισθολογική διαφορά. Είχαμε πρόσφατα την Ευρωπαϊκή ημέρα για την μισθολογική ισότητα ε, και απεδείχθη ότι οι γυναίκες, ε, ο μισθός των γυναικών είναι κατά 17,5% ε, χαμηλότερος για τις ίδιες επαγγελματικέ υπηρεσίες. Δεν υπάρχει δηλαδή ίση αμοιβή για την ίδια δουλειά ανάμεσα. celebrare la giornata Δεν υπάρχει λοιπόν ε, ακόμη η επιθυμητή ε, ισότητα ε, και οι γυναίκες χρειάζονται 14 μήνες σε κάθε χρόνο για να ε, έχουν τις ίδιες αποδοχές ε, ε, που έχουν οι άντρες σε διάστημα 12 μήνων. Γι' αυτό αποφασίσαμε να ιδρύσουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα της μισθολογικής ισότητας, διότι οι γυναίκες χρειάζονται δύο μήνες παραπάνω για να φτάσουν τον μισθό ε, των ανδρών. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μας απασχολεί όλους και θα ήθελα να συνυπολογίσετε και άλλα δύο στοιχεία, ότι ε, καλούνται να υπομιστούν ε, οι γυναίκες σε επιπρόσθετες ευθύνες, δηλαδή μεταξύ άλλων συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής. Δυστυχώς, Ο στόχος της συμφιλίωσης ε, της ε, προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Οι γυναίκες ε, ασχολούνται όχι μόνο με τα, τη φροντίδα των παιδιών, αλλά και τη φροντίδα των ηλικιωμένων ή των ασθενών μελών της οικογένειας, όχι απαραίτητα των ηλικιωμένων, τέλος πάντων ασχολούνται με την οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν ε, στον οικογενειακό πυρήνα. Οι γυναίκες λοιπόν έρχονται αντιμέτωπες ε, με μια ευρία γκάμα δυσκολιών και αποδεικνύεται ότι περιέρχονται σε ολοένα και πιο δεινή θέση οι γυναίκες αντί να βελτιώνεται η κατάσταση ε, η γυναίκα μην ξεχνάτε ότι δεν έχει πάτε τη δυνατότητα να έχει πλήρη απασχόληση. Όπως λέγαμε, χρειάζεται πολλές φορές να διακόψει την επαγγελματική της σταδιοδρομία για οικογενειακούς λόγους, για να ακολουθήσει το σύζυγό της ή για να φροντίσει τα παιδιά της. Ε, είναι δύσκολο λοιπόν ε, να συνταξιοδοτηθεί φυσιολογικά εφόσον ε, δεν έχει τον ίδιο αριθμό εισφορών, άρα ακόμη και εκεί εντοπίζεται ανισότητα, δηλαδή στην συνταξιοδότηση των ε, δύο φύλων. Θα ήθελα να προσθέσω ότι αν ασχοληθούμε με την ουσία του ζητήματος, αν παραδείγματος χάρη εξετάσουμε την κατάσταση με αριθμητικά στοιχεία θα συνειδητοποιήσουμε ότι ε, έχουμε περισσότερες πτυχιούχους από πτυχιούχους. Πάνω από 70% των πτυχιούχων στην Ευρώπη είναι ε, νέες γυναίκες που ε, είναι πιο έχουν ε, καλύτερη ε, επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά δυσκολεύονται παρόλα αυτά περισσότερο για να βρουν μια θέση απασχόλησης πέρα από τη διακεκομένη σταδιοδρομία ε, που αναφέραμε προηγουμένως. Προσπαθήσαμε στο δεύτερο ήμιση της ε, τωρινής θητείας να κάνουμε έναν απολογισμό. Συνειδητοποιείται ότι πληθυσμιακά υπερέχουν οι γυναίκες η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος είναι γυναίκες. Ε, εδώ στο Κοινοβούλιο όμως ε, οι βουλευτίνες ε, ανέρχονται στο 34% του συνόλου των βουλευτών. Σε σχέση με τις αντιπροέδρους, κυρία Κοκμέριν, κυρία Κράτσα, είναι αντιπρόεδροι. Έξι από τους 14, έξι από, ήταν ε, αντιπρόεδροι, συγγνώμη, έξι από τους 14 αντιπροέδρους ε, ήταν γυναίκες. Τώρα όμως ε, τρεις μόνο από τους 14 αντιπροέδρους είναι γυναίκες με τα νέα δεδομένα. Υπήρξε μεγάλη μείωση. Το ίδιο ισχύει και σε επίπεδο προέδρων και αντιπροέδρων των επιτροπών. Ε, σε επίπεδο Προέδρου Επιτροπών και Υποεπιτροπών από 24 ε, Προέδρους και Αντιπροέδρους μόνο 8 είναι γυναίκες. Ας πάρουμε τώρα τους υπαλλήλους. 3.000 είναι οι υπάλληλοι ε, στο Κοινοβούλιο, 58,8% είναι οι γυναίκες, όμως οι τμήματάρχες, γυναίκες τμήματάρχες αντιπροσωπεύουν ένα πολύ χαμηλότερο ποσοστό ε, είναι πασιφανές ότι εκτιμούνται οι επαγγελματικές δεξιότητες των γυναικών, όμως το οργανόγραμμα, οι ψηλότερες θέσεις παραμένουν ε, ακόμη στα χέρια των ανδρών. Επίσης έχουμε τις γυναίκες που υπήρξαν πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύο συγκεκριμένα, Δεν αρκεί φυσικά ε, σε ολόκληρη την ιστορία του Κοινοβουλίου να έχουμε μόνο δύο γυναίκες ε, προέδρους. Για να κλείσω την παρέμβασή μου, θέλω να τονίσω ότι είναι σημαντικό που έχουμε την θέληση να σημειωθεί πρόοδος και επίσης θα ήθελα να απευθύνω και ένα μήνυμα προς ε, τις νέες ε, συναδέλφους, ε, το κίνημα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών ε, δεν μπορεί να περάσει αποκλειστικά και μόνο μέσα από νομοθετικές πρωτοβουλίες. Παρότι χρειάζονται και τέτοιου είδους αποφάσεις, το βασικότερο είναι να αλλάξει η νοοτροπία μας. Ευχαριστώ πολύ Ρομπέρτα. Με πάθος παρουσίασες αυτό το θέμα, έκανες μια ζεστή εισαγωγή αναφέροντας τις προκλήσεις ε, τις οποίες αντιμετωπίζουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι οποίες φυσικά θα αντιμετωπίσουμε και για την επόμενη θητεία. Λοιπόν, ξέρουμε ότι δεν θα μας εγκαταλείψουν το πεδίο εύκολα αυτοί που το κατέχουν. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το κοινό μας που αποτελείται κυρίως από δημοσιογράφους θα πρέπει να μπορέσει να πάρει το λόγο. Έχουμε, νομίζω, εδώ στην αίθουσα όλους αυτούς που θα συμμετάσχουν στο πρώτο πάνελ. Ελάτε ε, εδώ να πάρετε θέση στο βήμα. Okay. So, dann beginnen wir. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρία Μπέρες. Δεν είναι ακόμα εδώ, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση αυτών που είναι εδώ. Ξέρετε ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο καθένας μπορεί να μιλήσει τη μητρική του γλώσσα. Και αυτό μας βοηθάει στην πολυμορφία. Ωραία. Είμαστε πλήρες στη σύνθεση του πάνελ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την παρουσίαση των μελών του πάνελ μας και θα ήθελα να σας πω από την αρχή ότι θα πρέπει να είμαι αυστηρή όσον αφορά την οργάνωση των συζητήσεων. Πέντε λεπτά για τα εισαγωγικά ε, σχόλια, την παρουσίαση και κατόπιν ερωτήσεις. Βεβαίως ε, το μικρόφωνο σας παρακαλώ πολύ να μην το μονοπολεί κανείς, ε, να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τους κανόνες της συζήτησης. Θα δώσω αμέσω το λόγο στην Περβόνς Περές. Μια γυναίκα με μεγάλη, θα έλεγα, και σημαντική επιρροή εδώ στα τεκτενόμενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με γνώσεις, με εμπειρογνωμοσύνη και όταν παίρνει το λόγο στην Ολομέλεια, ακούγεται. Είναι Γαλλίδα, ανήκει στο κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών και θα έλεγα ότι μας έχει συνηθίσει σε παθιασμένες παρεμβάσεις η Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου στα αριστερά μου ήταν στη θέση μου πριν από εμένα δηλαδή επικεφαλής της σημαντικής ομάδας που προεδρεύω μετά από εκείνην και φυσικά υπεύθυνη για θέματα επικοινωνίας. Είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία, όπως ξέρετε, γιατί η ισότητα των φίλων, οι ίσες ευκαιρίες, η έλλειψη διακρίσεων και η επικοινωνία είναι κάτι που κανονικά θα πρέπει να μας απασχολούν ταυτόχρονα. Με πολύ τολμηρές θέσεις για τα θέματα που μας αφορούν, ε, η κυρία Κράτα Τσαγκαροπούλη θα μας παρουσιάσει τις απόψεις της. Είναι Ελληνίδα και βεβαίως η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία όλα αυτά τα θέματα συζητούνται με πολύ ε, πάθος. Και βεβαίως Έχω εδώ και την την κυρία Οβίρη, η οποία η ίδια είναι γνώστη των θεμάτων αυτών, έχει τρεις κόρες, θα μας μιλήσει για την δική της εμπειρία. Η Μάργκιτ Κορνέλισεν των Πρασίνων από την Ολλανδία, μέλος της Επιτροπής Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι συντονίστρια των ε, Πρασίνων και υπεύθυνη για συζητήσεις και διαπραγματεύσεις μεταξύ της ομάδας, της πολιτικής ομάδας των Πρασίνων και άλλων ομάδων είναι αρμόδια για πολλά σημαντικά θέματα, μεταξύ των οποίων και τα θέματα των γυναικών. Έχουμε και ένα κύριο, τον κύριο Ντορνέα, ο οποίος είναι διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα ισότητας ευκαιριών. Και βεβαίως γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις προτάσεις που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα που αφορούν ε, την ίση μεταχείριση των γυναικών, τις θέσεις ε, που ανήκουν στις γυναίκες και προτάσεις για ε, το πώς θα μπορούσαμε να προωθήσουμε κάποιες δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Η κυρία Μπέρες θα πάρει το λόγο καταρχήν. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε μία εκπομπή που ήμουν καλεσμένη με ρώτησαν «Είστε υπέρ της κατάργησης της ημέρας των γυναικών» Απάντησα όχι βέβαια. Όχι επειδή ε, θα ήθελα ε, να καταργηθεί αυτή η ημέρα, αλλά δυστυχώς ξέρετε, ε, είναι πολύ νωρίς, είναι προώρο, δηλαδή χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν σήμερα να συζητήσουμε για αυτό το θέμα της ίσης αμοιβή. Δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει, να γίνεται αυτή η συζήτηση. Η Επιτροπή των Γυναικών είχε ήδη προτείνει να αναλυφθεί πρωτοβουλία ε, και αρνήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω τελευταία φορά να συνεδριάζουμε για ακριβώ το ίδιο θέμα. Μα είναι πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Έρχομαι από, προέρχομαι από μια χώρα όπου έχει λειτουργήσει το σύστημα της, ε, των οροσύμων του benchmarking ε, και για το θέμα της ισότητας ε, των δύο φύλων. Ε, παρόλα αυτά έχω την εντύπωση ότι δίνουμε τις μάχες μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί μιας κάκης της βάσης. Ποια είναι η εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι ότι με κατά έτσι. Προτείνεται να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ε, και καλύτερο είναι να ρυθμιστεί νομοθετικά το θέμα, διότι όλοι μιλάνε για την αυτορύθμιση. Να τι έχει γίνει στο, σε ολόκληρο τον κόσμο με την αυτορύθμιση αυτορύθμιση. Οπότε καλό θα ήταν ορισμένες φορές να χρησιμοποιούμε το νομοθετικό εργαλείο και τις ποσοστώσεις για να βελτιώσουμε την κατάσταση στην αγορά. Όμως δεν επαρκεί αυτό, δεν επαρκεί και ελοχεύει και ένας άλλος κίνδυνος ε, ότι είναι μια πρόταση θα την πω ε, γκλαμουράτη. Ε, ακούγεται πολύ ωραία α, γιατί θα ρυθμίσει τα ζητήματα, λένε, της διοίκησης των επιχειρήσεων και τα Δεν ισχύουν αυτά δηλαδή. Στο ε, το... Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι κέριο το ζήτημα όχι μόνο για τις γυναίκες αλλά και για όλες οι υπόλοιπες ε, πληθυσμιακές ομάδες. Στην Επιτροπή Γυναικών ε, είναι γνωστά όλα αυτά. Αγωνιζόμαστε, κινητοποιούμαστε, χρησιμοποιούμε διάφορα νομοθετικά εργαλεία για την, να επιτύχουμε την ίση ομοιβή, την ισότητα των ε, γυναικών με τους άντρες. Εάν λοιπόν κερδίσουμε αυτές τις μάχες θα έχουμε κάνει κάτι συγκεκριμένο, ούτως ώστε να αναβιώσει ε, το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο που ε, δυστυχώς πνέει τα λίστια. Δεν θέλω να υπερβώ και το χρόνο μου, θα κλείσω σε λίγο. Ασχολούμαστε λοιπόν με τα θέματα των γυναικών, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται για ζητήμα των πολιτών. Και δεν μου βγαίνει από το μυαλό αυτό που συνέβη στο Αφγανιστάν. Θυμάστε, εμείς ήμασταν εδώ στο Κοινοβούλιο κινητοποιημένοι, ενώ φορούν φορούσαν ε, ολόζωμη μπουρκα στο γυναίκες ε, στο Αφγανιστάν ε, και κανείς δεν ήθελε να ασχοληθεί με αυτό μέχρι που αποφάσισαν να στείλουν το στρατό και τα όπλα και τότε συνειδητοποίησαν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ε, πολιτικά αντικειμενική θεώρηση των πραγμάτων, να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση. Νομίζω ότι πρέπει να αγωνιστούμε για την ισότητα, για το καλό και των γυναικών και των ανδρών. Χαίρομαι που αναλαμβάνεται και πάλι η πρωτοβουλία από το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω κάποιο να δώσει την όθηση που χρειάζεται σε αυτό το θέμα. Σα ευχαριστούμε κυρία Μπερέ, ε, κυρία Κόχ, για αυτήν την σύντομη εισαγωγή και τα βασικά σημεία τα οποία τονίσατε στην παρέμβασή σα, Δεν περιμένουμε άλλο. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κράτσα Τσαγκαροπούλ, παρακαλώ. Merci beaucoup, madame. Euh, Ευχαριστώ πολύ την συντονίστρια. Θα ήθελα να εκφράσω την μεγάλη ικανοποίησή μου που βρίσκομαι ενώπιον σε σήμερα σε αυτό το ετήσιο ε, ραντεβού μας ε, με τους εταίρους ε, της κοινωνίας των πολιτών και όλος ιδιαιτέρως του τύπου ούτως ώστε να συζητήσουμε για αυτά τα τόσο βασικά ζητήματα του ρόλου της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία, της ισότητας, της αμοιβή και όλων των ε, πρωτοβολιών και των εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ημέρα των γυναικών. Να συγχαρώ και πάλι τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ε, ε, που πριν από δύο μήνες ήταν υπό τη δική μου ευθύνη. Ευχαριστούμε επίσης την υπηρεσία τύπου που μας δίνει κάθε χρόνο αυτή την ευκαιρία. Θα συνεχίσω στα ελληνικά. Ε, tout ναι, ότι μπορούμε να να μοιραστούμε μαζί μια διαπίστωση, στην οποία αναφέρθηκε και μόλις και η κυρία Περβόνσο Περές, ότι το φαινόμενο αυτό της ανισότητας που μας καλεί να διατηρούμε την Παγκόσμια ημέρα α, της γυναίκας, την 8η Μαρτίου, είναι ένα φαινόμενο και παγκόσμιο και διαχρονικό. Και πρέπει κάθε χρονιά, τέτοια μέρα ιδιαίτερα, να διαρωτηθούμε όλοι μαζί γιατί παρόλη τη συνειδητοποίηση που υπάρχει σήμερα τη σημασία που έχουν οι ανισότητες γιατί επιμένει η ανισότητα στην κοινωνία μας τόσο στον ανεπτυγμένο κόσμο όσο και στον κόσμο φυσικά που προσπαθεί να περάσει σε μια φάση ε, δημοκρατικής διακυβέρνησης. Και τα στερεότυπα και οι αντιστάσεις επιμένουν. Οπότε εμάς σαν πολιτικούς και σας σαν δημοσιογράφους μας καλεί ιδιαίτερα αυτή η διαπίστωση να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο έργο μας. Διότι και τα στερεότυπα και οι αντιστάσεις έχουν ανάγκη από σωστές πολιτικές, αλλά και από ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, εγρήγορση της κοινή γνώμης, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως από τις συναδέλφους μας. Είναι, πιστεύω, ένα μήνυμα και μια δέσμευση που πρέπει να πάρουμε στο τέλος αυτής της ημέρας. Ερχόμενοι μετά στο θέμα της ε, Παγκόσμιας ημέρας, της φετινής και γύρω από το οποίο ε, ε, γίνεται και το σημερινό σεμινάριο, η διαφορά αμοιβών. Είναι σκανδαλώδες μετά το να έχουμε ακόμη αυτό το θέμα προς αφού και στα συντάγματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγράφεται η ανάγκη ίσων αμοιβών και είναι και θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πρώτη, από το, τη, τη, την πρώτη συνθήκη της ε, Ρώμης το 1957. Πιστεύω ότι έχει δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος. Απ' τη μια μεριά οι ανισότητες της αμοιβέ εκφράζουν τις ανισότητες των δύο φίλων στην κοινωνία, παράλληλα η συνέχιση των ανισοτήτων στις αμοιβέ ενισχύουν την ανισότητα των δύο φύλων στην επαγγελματική δραστηριοποίηση, στην ανέλυξη, στην σταδιοδρομία, στην επίτευξη στόχων, διότι η, η, η, η ανισότητα στις αμοιβέ δηλώνει ότι οι γυναίκες δεν είναι ενδυνάμοι, εργαζόμενες ε, ε, για υψηλά πόστα, για, μεγάλες, ε, ε, για μεγάλη αξιοποίηση όπως είναι οι άνδρες. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει να αποτελεί το θέμα της καμπάνιας μας σήμερα, διότι έχει γίνει ένας φαύλος κύκλος γύρω από αυτό στην κοινωνία μας. Αυτό το οποίο θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ, που έχει να κάνει και με την έκθεση την οποία έχω επιβάλει και έχει ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι η ανισότητα στην ανέλυξη, η δυσκολία να φτάσουν οι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, έχει για μένα μια συμβολική και ουσιαστική σημασία, συμβολική διότι η ανέλυξη των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια σημαίνει ότι μπορεί να σπάσει άλλη οροφή και ουσιαστική διότι πιστεύουμε ότι αυτό θα επιφέρει ε, καλύτερα αποτελέσματα οικονομικά τόσο στην ε, επιχείρηση τόσο και στην οικονομία και την κοινωνία μας ευρύτερα, όπως μας δείχνουν όλες οι μελέτες. Απαντώντας λοιπόν, κυρία Συντονίστρια, στο θέμα του πάνελ το οποίο μα θέσατε προς συζήτηση, πώς η ανισότητα αμοιβών επηρεάζει την ανάπτυξη και το προϊόν, το ακαθάριστο προϊόν της κοινωνίας και της οικονομίας μας, θα σας έλεγα ναι, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουμε στη διάθεσή μας. Υπάρχουν μελέτες που είναι πολύ τολμηρές, που μας λένε ότι αν καλύψουμε το μισθολογικό χάσμα θα έχει θεαματικά αποτελέσματα η επιχείρηση. Διότι σημαίνει ότι οι γυναίκες θα αξιοποιηθούν, θα αναβαθμιστούν και θα δώσουν όλα αυτά τα χαρίσματα, τα έμφυτα και τη, της τα αποκτήματα τα οποία τα χάνει η επιχείρηση σήμερα. Ε, είναι κάτι στο οποίο βασίζεται και η έκθεση η οποία συνέταξα και ψηφίστηκε, τη σημασία που έχει για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή η επίτευξη της μισθολογικής ισορροπίας. Δεύτερον, κάτι παράδοξο το οποίο ε, διεπίστωσα ε, κάνοντας την έρευνα για την έκθεσή μου. Η ίδια διαφορά μισθολογική υφίσταται και στις υψηλές θέσεις. Εγώ πίστευα ότι η διαφορά μισθολογική είναι στις θέσεις τις χαμηλές. Εκεί που οι γυναίκες μπαίνουν στην αγορά εργασίας χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις, λόγω στερεοτύπων, λόγω υποχρεώσεων οικογενειακών, λόγω φιλοδοξίας και δέσμευσης να, να φτάσουν ψηλά, αλλά μια και φτάνουν σε, ψηλά επίπεδα δεν υπάρχει πια το θέμα της μισολογικής διαφοράς. Το θέμα της μισολογική διαφοράς λοιπόν υπάρχει στα υψηλά επίπεδα, κάτι που συνεχίζει να εκφράζει τις ανισότητες στην κοινωνία και παράλληλα στέλνει ένα πολύ αρνητικό μήνυμα ότι μια γυναίκα που κατάφερε με τις δυσκολίες που έχουν οι γυναίκες σήμερα να χτίσει μια καριέρα στον πολύ απαιτητικό και ανταγωνιστικό ιδιωτικό τομέα να φτάσει σε μια θέση ε, senior, σε μια executive θέση σε ένα διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να είναι θύμα των στερεοτύπων και να έχει ε, το δικαίωμα η επιχείρηση, ο εργοδότης να την ανταμείβει λιγότερο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να, συνε... συνειδητοποιήσουμε ότι τα στερεότυπα αυτά και αντιστάσεις ακολουθούν τις γυναίκες σε όλα τα επίπεδα, μετά από οποιαδήποτε προσπάθεια καριέρας και ότι υπάρχουν χώρες που γίνεται μια συζήτηση σοβαρή, λαμβάνονται τέτοια νομοθετικά μέτρα, παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, πρόσφατα και στην Ιταλία υπάρχουν και χώρες και εδώ έρχομαι σε κάτι που είπατε, δεν συμφωνώ μαζί σας ότι σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα γίνεται αυτή η συζήτηση και εδώ φέρνω τη χώρα μου σαν παράδειγμα, λόγω των μεγάλων δημοσιονομικών προβλημάτων που έχει υπάρχει η, επικρατούσα άποψη ότι έχουμε άλλα προβλήματα να λύσουμε και μετά τα θέματα της ισότητας. Προσπάθεια και αγώνας μας είναι να εντάξουμε την ισότητα και στην ανάπτυξη και στη δημοσιονομική προσαρμογή διότι οι γυναίκες είναι πολύτιμα αγαθά που τα έχει ανάγκη η Ευρώπη είτε για να καλύψει τα ελλείμματα τα δημοσιονομικά είτε για να κάνει το αναπτυξιακό της άλμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ähm, Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι Πραγματικά τα θέματα που έχουμε θέσει σε αυτό το πάνελ, σε αυτή τη ζήτηση είναι πολλά και μπορούν να συζητηθούν από πολλές ε, πτυχές. Η κυρία Ρέντινγκ έχει κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχει η έκθεση με πολύ πλούσιο ε, περιεχόμενο. Έχουμε και πιο ριζοσπαστικές ε, προτάσεις που θα μπορούσαμε να προωθήσουμε. Θα δώσω το λόγο όμως στην ε, επόμενη ομιλήτρια, Θηριόβιν, και κατόπιν ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε και στις ε, ερωτήσεις και απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι από την Εστονία. Σήμερα που συζητούμε για την ίση αμοιβή η συνεργασία, οφείλω να παραδεχθώ ότι ντρέπομαι. Ντρέπομαι γιατί είμαστε ουραγοί, είμαστε πολύ κακοί μαθητές. 30% είναι το μισθολογικό χάσμα στη χώρα μας. Και ο φορέας τον οποίο εκπροσωπώ έχει επομένως ασχοληθεί με το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών στη χώρα μας. Πάντως, είναι και το θέμα των ε, ατομικών ελευθεριών, είναι το θέμα της ισότητας γενικότερα. Και το θέμα δεν είναι μόνο μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όλοι, όλες οι κοινωνικές ομάδες ε, δικαιούνται ε, την ισότητα. Θέλουμε επομένω να καταφέρουμε να έχουμε τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες και στο χώρο εργασία. Σε οποιαδήποτε θέση στην ιεραρχία κάποιας ε, εταιρείας. Εμείς στο Σύνταγμα μας έχουμε κατοχυρώσει την αρχή της ισότητας του Σύνταγμα και σε άλλους νόμους του κράτους. Το 1957 με την ε, συνθήκη της Ρώμης κατοχυρώθηκε και εκεί η αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία. Όμως, να που σήμερα το 2012 ακόμη αυτά τα συζητάμε. Το 2008 πάντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση της κυρίας Μπάουερ που αφορούσε ακριβώς το σημερινό μας θέμα. Από το έχουν περάσει τέσσερα χρόνια, όμως σημαντική μεταβολή δεν έχει σημειωθεί. Δεν ε, πρέπει να κατηγορούμε μόνο την ε, χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν είναι μια τέτοια σωστή προσέγγιση. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι θα πρέπει να αναλάβουμε δράση, ότι θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και θα πρέπει να γεφυρωθεί αυτό το μισθολογικό χάσμα, το οποίο βέβαια οφείλεται σε ένα σωρό παράγοντες. Σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα δυσμενή για τις γυναίκες στερεότυπα. Αυτό βέβαια παίρνει χρόνο. Έτσι να καταφέρουμε αυτές οι αρχές που εδώ και 40 χρόνια διατυπώθηκαν και κατοχυρώθηκαν να υλοποιηθούν. Υπάρχουν στατιστικά δεδομένα. Η Eurostat συλλέγει τα δεδομένα και καταρτίζει τους πίνακές της. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσον τα δεδομένα που αφορούν την ε, αμοιβή για την εργασία κατά πόσον λέω είναι ακριβή τα δεδομένα διότι πολλές φορές τα δεδομένα που συλλέγει ο Ροστάτ από πολλούς κλάδους είναι στοιχεία που αφορούν μόνο τους άντρες. Έτσι επομένως δεν μπορούμε να έχουμε συγκρισιμότητα. πάνω από τις μισές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θεσπίσει νομοθετήματα για την ισότητα. Και αυτές οι χώρες έχουν συγκρίνει τα δεδομένα για τις αμοιβέ, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε όλες τις χώρες. Άρα χρειάζεται περισσότερος κοινωνικός διάλογος και χρειάζεται με κάποιο τρόπο γύρω στο να μπορεί να συλλέξει αντικειμενικά δεδομένα που να αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση. Για την πολιτική ομάδα των φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγώ έχω διατελέσει συγκίτρια, σκηνώδες συγκίτρια, έχω προτείνει τροπολογίε για τις εκθέσεις που αφορούν το ζήτημα τούτο και έχουμε την έκκληση σε όλες τις χώρες να μπορέσουν με <clears throat> δεσμευτικό τρόπο να συλλέξουν και να αναλύσουν τα δεδομένα που σας είπα. Και γι' αυτό και ελπίζουμε ότι σε λίγα χρόνια που θα ξαναχρειαστεί να τα πούμε, τότε ελπίζουμε να έχουν σημειωθεί κάποιες αλλαγές, προς το καλύτερο βέβαια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σύρι Και ιδιαίτερα γιατί αναφέρθηκε σε κάποια πιο μελανά σημεία στη δική σου χώρα. Βεβαίως, μιλάμε συχνά για τους μέσους όρους ε, στην Ευρώπη, αλλά οι διαφορές συνεχίζουν να είναι πολύ σημαντικές από τη μια χώρα στην άλλη στους διάφορους τομείς. Θα συνεχίσουμε όμως με την Μαρή Κονέλισεν πέντε λεπτά και όχι παραπάνω. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που είστε τόσο πολύ εδώ στην αίθουσα. Το θέμα είναι σημαντικό και το χάσμα το μισθολογικό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα γιατί ουσιαστικά προσθέτει ακόμα μία ανισότητα στην αγορά εργασίας. Και βεβαίως υπάρχουν ε, τα λεγόμενα προσαρμοσμένα και μη προσαρμοσμένα χάσματα μεταξύ των μισθών και των αποδοχών ανδρών και γυναικών. Ένα σύνολο διακρίσεων χαρακτηρίζουν αν θέλετε, τις ε, αποδοχές ε, των ανδρών και των γυναικών και πολλές φορές μιλάμε για προσαρμοσμένα στοιχεία που ουσιαστικά ενσωματώνουν το σύνολο των ε, ανισοτήτων. Παραδείγματος χάρη, διαφορετικές ε, συμβάσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένας άνδρας και μια γυναίκα ε, πληρώνονται διαφορετικά, οι γυναίκες πληρώνονται λιγότερο για μία ώρα εργασίας, αντίστοιχης εργασίας. Πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσει κανείς αυτές τις διαφορές. Πολλές φορές αυτές οι διαφορές και ανισότητες αυξάνονται με τα χρόνια και κατά τη διάρκεια ε, της σταδιοδρομίας. Επίσης ε, αυτές οι ανισότητες και διαφορές είναι δύσκολο να εντοπιστούν αυξήθηκαν επίσης με την κρίση. Αυτό βέβαια δεν φαίνεται ακόμα στα στοιχεία που διαθέτουμε. Είναι πολύ νωρίς για να υπολογιστούν. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία δείχνουν τις ανισότητες όπως επιδόματα, έλλειψη αποζημιώσεων ε, για ό,τι έχει σχέση με τις επιπλέον δραστηριότητε που έχουν οι γυναίκες, οι διακοπή των επαγγελματικών σταδιοδρομιών, τα ανώτατα όρια, οι λιγότερες προσφορές ε, όσον αφορά τις γυναίκες, επαγγελματικές ευκαιρίες. Όλα αυτά αυξάνουν τα χάσματα, τα μισθολογικά. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι οι αριθμοί δεν είναι σωστοί. Πολλές φορές ε, στα χαρτιά τα χάσματα μεταξύ των μισθών των ανδρών των γυναικών εμφανίζονται πολύ μικρότερα. Λιγότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι, αν θέλετε, ένα φαινόμενο το οποίο ουσιαστικά μειώνει τις διαφορές. Γι' αυτό και, παραδείγματο χάρη στην αγορά εργασίας της Πολωνίας, τα πράγματα φαίνονται ρόδινα. Ελάχιστες γυναίκες όμως βρίσκονται σε αυτήν την ε, αγορά εργασίας της Πολωνίας. Γι' αυτό και η κατάσταση φαίνεται τόσο θετική. Η πραγματικότητα λοιπόν πολλές φορές θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια πιο προσεκτική παρακολούθηση της κατάστασης έτσι ώστε να μπορέσουμε να διακρίνουμε αυτές τις ε, διαφορές. Όπως παραδείγματο χάνει τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα με τον φόρο αλληλεγγύη και το πώ αυτό αντικατοπτρίζει ε, τη διαφορετική αντιμετώπιση και το διαφορετικό βάρος που θα επομιστούν οι άνδρες και οι γυναίκες. Αυτό που πολλές φορές βλέπουμε είναι ότι αν, μια γυ... αν ε, ένας κλάδος επαγγελματικός ξαφνικά αποκτήσει περισσότερες γυναίκες από ότι άνδρες, ξαφνικά υποβαθμίζεται. Το ίδιο έγινε με πολλούς επαγγελματικού κλάδους, όπως παραδείγματο χάρη η δάσκαλη που ήταν καθαρά ανδρικό επάγγελμα, σήμερα έχει γίνει γυναικείο επάγγελμα και την ίδια ώρα έχει υποβαθμιστεί από όλες τις απόψεις και όσον αφορά βεβαίως τις αποδοχές άδειες μητρότητας. Οι γονικέ άδειε. συνεχίζουμε να τις ονομάζουμε άδειες μητρότητας, διότι βεβαίως πολύ περισσότερες γυναίκες ε, ζητούν και παίρνουν αυτές τις άδειες. Θα ήταν πολύ καλό κάποια από τα μέτρα που σήμερα υποστηρίζουν και βοηθούν τις γυναίκες να γίνουν δεσμευτικά, δεσμευτικά για όλους τους εργοδότες. Επαναλαμβάνω, οι διαφορετικές συμβάσεις συνεχίζουν να κρύβουν την πραγματικότητα διαφορετικές συμβάσεις εργασίας, άτυπες συμβάσεις εργασίας. Ξέρετε, ότι εμείς ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε το θέμα του Στρασβούργου και βεβαίως την ε, ανάθεση της φροντίδας των παιδιών κατά τη διάρκεια αυτών των μετακινήσεων. Έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία έτσι ώστε να υπάρξουν συνεργαστικά μέτρα για την μετακίνηση του Στρασβούργου. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να πάνε να κοιμηθούν στο Στρασβούργο χωρίς ε, τα παιδιά. Ε, ξέρετε και εγώ πρόσφατα έκανα παιδί και μπορώ να σας καταλάβω όταν τα λέτε αυτά. Πέρα από τα αστεία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, για τα στοιχεία που μας δώσατε, για τις διάφορες κατηγορίες ε, και σε πέντε λεπτά μπορείτε να μας πείτε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για ε, τα θέματα των, ε, της ισότητας των δικαιωμάτων γυναικών και των αντρών, ο κύριος Σομπάνου Ντορντέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, αξιότιμα μέλη, αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή ευκαιρία που μας δίνετε ενώπιον των δημοσιογράφων να σας εξηγήσουμε, δηλαδή ποιες προσπάθειες καταβάλουμε για να επιτύχουμε ακριβώς ε, τον ίδιο στόχο που εκθέσατε κι εσείς ε, λεπτομερώς ε, στις παρουσιάσεις σας. Πρόκειται για μια πάρα πολύ θετική πρωτοβουλία που αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση του κοινού μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία που έχει αυτό το ζήτημα. Αναφέρθηκατε ε, στην ίση αμοιβή για ίση δουλειά είναι μια αρχή που προβλέπεται ε, στις ε, συνθήκες από το 57, δηλαδή από τις ιδρυτικές συνθήκες της τότε ΟΚ. Παρόλα αυτά, σήμερα παρατηρούμε ε, ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα και αυτό δεν οφείλεται τόσο πολύ στις άμεσες διακρίσεις ε, αλλά κυρίως στις συνθήκες της αγοράς όπου εξακολουθεί να παρατηρείται αυτή η μισθολογική διαφορά. Είναι ένας ιδιαίτερα αποθαρρυντικός για τις γυναίκες παράγοντες σχετικά με την είσοδό τους ή την ε, ε, εκ νέου είσοδο μετά από μία διακοπή στην ε, αγορά εργασίας. Επλήττονται επίσης οι οικονομίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι κοινωνίες των ε, ε, κρατών της Ένωσης. Επηρεάζονται επίσης δείκτες της κοινωνικής ανάπτυξης ε, και ούτε καθεξής. Οπότε θα ήθελα να σας πω ότι συστηματικά πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση, όχι μόνο άπαξ το χρόνο όταν εορτάζουμε την ημέρα, την Ευρωπαϊκή ημέρα της Ισαμβής, όπως την περασμένη εβδομάδα, παραδείγματος χάρη, πάγια θα πρέπει να λαμβάνουμε δεόντως υπόψη αυτό το ζήτημα σε όλες τις δράσεις μας. Με ρωτήσατε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει σε δύο επίπεδα να αναλυφθεί η δράση πρώτον, πρέπει να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση όχι μόνο της κοινή γνώμης αλλά και των οργανώσεων εργοδοτών, των ίδιων των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των ίδιων των εργαζομένων ε, για την ύπαρξη αυτού του πελώριου χάσματος, λαμβάνοντας υπόψη τις, ε, κρατικές ιδιαιτε... τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, κάθε χώρα έχει ε, ρυθμίσει με συγκεκριμένο τρόπο την αγορά εργασίας όπως παρα... και ρυθμίζει θέματα όπως ο μισθός, παραδείγματο χάρη. Σε ορισμένες χώρες αυτό είναι αντικείμενο συλλογικών ή επιχειρησιακών συμβάσεων, σε άλλα κράτη είναι νομοθετικό το ζήτημα. Γνωρίζουμε ότι στις χώρες όπου όπου νόμοθετικός ρυθμίζεται η αμοιβή, το χάσμα αυτό είναι κάπως μικρότερο σε σχέση με τα κράτη-μέλη όπου ο μισθός ορίζεται ε, κατά ε, γενικό λόγο μετά από ε, συλλογικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις. Οπότε θα πρέπει να βελτιώσουμε την ευαισθητοποίηση του, της κοινή γνώμης για την ύπαρξη αυτής της διαφοράς και να αποταθούμε στους βασικούς εταίρους, βασικούς παίκτες που επηρεάζουν την κατάσταση. Επίσης, θα πρέπει να αποδώσουμε σημασία στην νομοθετική διάσταση. Με την αρχή αυτή όμως που προβλέπεται στις ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έλεγα ότι είμαστε σχετικά ασφαλείς νομοθετικός πόρτ. Δηλαδή, έχουμε την οδηγία το 2006, αναθεωρημένη οδηγία συγκεκριμένα, που έχει ως αντικείμενο είναι ίση μεταχείριση των γυναικών και άνδρων στον χώρο εργασίας τους. Πρόκειται για μια αναθεωρημένη οδηγία, όπερ σημαίνει ότι εγκρίθηκε πρώτου 2006 η οδηγία. Αυτό καλύπτει το ζήτημα της άμεσης και έμεσης διακριτικής μεταχείρισης ε, που παρατηρείται. Γι' αυτό το λόγο πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να διοικητεύσουμε τις προσπάθειές μας κυρίως ε, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των κοινωνικών εταίρων αλλά και των μεμονωμένων ατόμων σχετικά με την ύπαρξη αυτού του μισθολογικού χάσματος. Γι' αυτό το λόγο πέρσι για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανώσαμε ε, ε, μια παρουσίαση για το θέμα αυτό ε, ευκαιρία τη ημέρα τη μισθολογική ισότητα. Ε, δεύτερη φορά συμβαίνει αυτό φέτος. Έχουμε από το 2010 μια συγκεκριμένη στρατηγική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το ίδιο ζήτημα, εντατικές ενημερωτικές εκστρατείες που απευθύνονται μεταξύ άλλων και στο κοινό. Σας δείχνω τώρα αυτή τη στιγμή τα πρόσωπα αυτής της εκστρατείας που πρέπει να συνειδητοποιήσετε ε, ότι τα πρόσωπα που χρησιμοποιούμε θα πρέπει να ταιριάζουν στον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και στην κοινωνία. Δηλαδή τους βασικούς αποδέκτες ε, του μηνύματος μας. Ε, βλέπετε αυτά τα πρόσωπα που εμφανίστηκαν στα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν περιοριστήκαμε σε αυτό. Πήγαμε επίση στα ίδια τα κράτη-μέλη για να συνομιλήσουμε και με τους εργοδότες και με τους εργαζόμενους. δημιουργήσαμε ιστοσελίδα δε σε 22 γλώσσες σχετικά με τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία και τα αίτια του μισθολογικού χάσματος. Ε, ε, συνδιοργανώσαμε εκδηλώσεις επιτόπου στα κράτη-μέλη για το ζήτημα αυτό. Τους καλέσαμε τα κράτη-μέλη να ε, συνεργαστούν μαζί μας για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής ημέρας της Μισθολογικής Ισότητας και τώρα οργανώνουμε μια εκστρατεία με αποδέκτες της επιχειρήσεις. Αρχίζει ήδη φέτος η εκστρατεία αυτή, δηλαδή θα συναντηθούμε με επιχειρήσεις ούτως ώστε να τους ενθαρρύνουμε και να προβούν σε ανταλλαγή ε, βέλθων πρακτικών ε, σχετικά με την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, εξάλλου η κυρία Πέγβανος Μπέρες ε, το προανέφερε, υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα που η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Βίβιαν Ρέντινγκ, ε, σχολίασε τη Δευτέρα ε, στην τηλεόραση. Καλούνται λοιπόν ε, μέλη διοικητικών συμβουλίων εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών και δεν είναι θέμα απλώς προβολής, γιατί το 2010 σας υπενθυμίζω ότι στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εδώ σας το δείχνω, πρόκειται για ένα δημόσιο έγγραφο που ε, πραγματεύεται το θέμα της συμμετοχής των γεργών, όχι μόνο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο επιχείρησης, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ δεν εισηγήθηκε κάτι συγκεκριμένο, προέβη απλώς στην παρουσίαση της έκθεσης που εκπονήσαμε και που βασίστηκε στα στοιχεία μιας δημόσιας διαβούλευσης που ξεκίνησε τη Δευτέρα και θα διαρκέσει τρεις μήνες σας καλούμε όλους να μετάσχετε σε αυτή τη διαβούλευση. Μετά το πέρας της διαβούλευσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει ε, την σχετική απόφαση. Σας ευχαριστούμε. Ε, δηλαδή νομοθεσία και ευαισθητοποίηση του κοινού είναι τα, οι δύο λέξεις κλειδιά της παρουσίασής σας. Νομίζω ότι η καταληκτική ε, πρόταση της ε, ομιλίας σας ε, έχει ιδιαίτερο βάρος. Θα ήθελα να ακούσουμε τώρα τα σχόλιά σας και Ελπίζω και πιστεύω ότι θα έχετε πάρα πολλές παρατηρήσεις, ε, ε, πάρα πολλά σχόλια. Ε, για κάποιον από όλους τους ομιλητές του πάνελ θα ήθελα τώρα να σας δώσω το λόγο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Εγώ έχω πάντως, αν δεν έχετε εσείς. Έχετε το λόγο, παρακαλούμε. Πέστε μας το όνομά σας πρώτα. Και πατήστε το κόκκινο κουμπάκι για το μικρόφωνο από τη Βιέννη. Η ερώτησή μου αφορά το έξη; Είπαμε πολλά για την ε, δικαιοσύνη, για τους νόμους, πώς μπορεί να θεσπιστεί η ισότητα όμως και η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να ωφεληθούν από όλα αυτά. Δηλαδή θέλω να σα πω τι μπορούμε να κάνουμε τόσο ώστε να δημιουργήσουμε ένα πλεονέκτημα για την οικονομία της επιχειρήσης, τη εταιρεία, τόσο ώστε και εκείνοι να έχουν κίνητρο να βοηθήσουν στην ισότητα. Γιατί δεν του νοιάζει άπαξ και κερδίζουν ε, τι γίνεται. Του αρκεί το να υπάρχει κέρδο. Άρα πώ θα δημιουργήσουμε κίνητρα πλεονεκτήματα για τη βιομηχανία, για την οικονομία, ώστε και εκείνοι να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει, χωρί να του υποχρεώνει κανένα να είναι δίκαιοι και σωστοί. Γιατί αυτό τους νοιάζει, δεν τους νοιάζει δικαιοσύνη, τους νοιάζει το κέρδος. Η ερώτησή σας απευθύνεται σε κάποιον συγκεκριμένα ή μπορεί να απαντήσει οποιοδήποτε από το πάνελ. Ποιος θα ήθελε το λόγο? Εγώ. Yeah. Um, it, it is definitely a... Οπωσδήποτε χρειάζεται και το καρότο και το ραβδί και τον μπαστούνι διότι δεν είναι τόσο εύκολο να ξεκαθαρίζει κανείς στην κάθε μία εταιρεία και επιχείρηση πόσο θα κερδίσει γιατί υπάρχουν βέβαια άπειρος αριθμός ερευνών που ξεκαθαρίζει το πόσο ωφελεί το να έχει κανένας πολλές γυναίκες σαν στελέχη ε, στην κορυφή της πυραμίδας εταιρείας και ότι είναι καλό αυτό για τις δουλειές Μιλάμε για 35% περισσότερο εισόδημα, περισσότερο, περισσότερα έσοδα. Όμως είναι δύσκολο αυτά τα οποία επί χρόνια κάνανε να τα αλλάξουν. Άρα χρειάζεται μπαστούνια. Χρειάζονται και οι Ρώσεις όσον αφορά τις δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος των ε, γυναικών όταν δηλαδή για την ίδια δουλειά αμείβονται λιγότερο. Επίσης, Χρειαζόμαστε και μέτρα για τη διαφάνεια. Να καταλάβουν οι εργοδότες ότι θα πρέπει να διακρίνει διαφάνεια το τι πληρώνουν. Να ξέρει δηλαδή ο κόσμος πόσο πληρώνεται, το οποίο δεν είναι πάντα αυτονόητο. Κοιτάξτε, εμεί τώρα είμαστε από διαφορετικά πολιτικά κόμματα, οπότε όταν κάτι λέει κάποιο, αυτό δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά και οι άλλοι το, το, το, το, το σπαζόμαστε. Εγώ βέβαια που είναι από τη συζήτηση πρέπει να είμαι ουδέτερη προέρχομαι από άλλη πολιτική ομάδα. Τέλο πάντων, τώρα θα ήθελα το λόγο, κύριε Κάτσα, που είναι, προέρχεται από του συντηρητικού. Ευχαριστώ πολύ. Ε, για το θέμα αυτό, ήθελα να σα πω ότι με την κυρία Κορνέλισεν, που μόλι μίλησε προηγουμένω, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία στο πλαίσιο τη έκθεση που συνέταξα και που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εκεί, παρόλο που το θέμα είναι οι γυναίκε στο leadership των επιχειρήσεων, και παρόλο που η πρότασή μας είναι πολύ συγκεκριμένη, Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν διαπιστώσει ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει εξέλιξη, πρέπει να προβεί σε νομοθετική πρωτοβουλία. Ε, αναδεικνύονται όλες οι προκλήσεις της ανέλυξης των γυναικών. Διότι ναι μεν, ε, όπως είπε και η κυρία Περβάνς Περές, ε, το να τοποθετήσουμε αυτόματα πολλές γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια μπορεί να θυμωρηθεί ότι είναι και μια γκλαμούρο ε, δράση δεν λύνει το πρόβλημα της κοινωνίας. Εμείς ζητούμε να αναδειχθούν οι γυναικείες ικανότητες ούτως ώστε να είναι αυτονόητο να φτάσουν οι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια διότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι εταιρείε αναζητούν γυναίκες και δεν βρίσκουν. Ενώ όλοι ξέρουμε πόσα ταλέντα υπάρχουν στην κοινωνία και στην οικονομία, αναζητούν και δεν βρίσκουν. Γι' αυτό η διαφάνεια, νέος τρόπος του management, η διευκόλυνση οικογενειακής και ε, επαγγελματικής ζωής, το mentoring, η παρακολούθηση της καριέρας ιδιαίτερης ιδιαίτερων περιπτώσεων γυναικών η διευκόλυνση της ε, κινητικότητας από μια χώρα στην άλλη βάσει των οικογενειακών υποχρεώσεων για τις γυναίκες είναι στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την φυσιολογική ανέλυξη των γυναικών στο management των επιχειρήσεων συν βέβαια την ευαισθητοποίηση και την πολιτική βούληση και των ε, ίδιων των ηθινόντων ε, στις επιχειρήσεις. Αλλά επανέρχομαι έτσι να συμπληρώσω ότι η πρότασή μας δεν είναι απλά πάρτε μια νομοθεσία για 40% των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, είναι ένα πακέτο συμπληρωματικών δράσεων που πρέπει να συνοδεύουν αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία που εμείς πιστεύουμε ότι την έχει ανάγκη η κοινωνία σαν ένα γεγονός που θα ανάψει, θα ξεκινήσει ε, μια νέα διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν και άλλα μέλη του πάνελ που θέλουν να απαντήσουν σε ερωτήσει σα, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Αν μπορείτε να απαντάτε σύντομα, το λέω απλώ για να μπορέσουμε να απαντήσουμε περισσότερες ερωτήσεις. λα, λα. Έλα. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να δούμε το πώς θα δείξουμε με τρόπο απτό, χειροπιαστό, το πόσο συμφέρει, το πόσο είναι καλό το να υπάρχει αυτή η ισότητα στην ε, αμοιβή. Πολλές φορές οι γυναίκες, τουλάχιστον αυτές στην Ευρώπη, είναι πιο καλά καταρτισμένες. Έχουν καλύτερες σπουδέ, περισσότερες δεξιότητε προσόντα από τους άντρε. Έχουμε ένα σωρό μελέτες που κατατείνουν σε αυτό. Και επίση προκύπτει αβίαστα ότι οι γυναίκε είναι πάρα πολύ καλέ στο να λαμβάνουν αποφάσει. Και όσο πιο ψηλό επίπεδο κάποιε εταιρείε λαμβάνουν αποφάσει από γυναίκε, τόσο πιο μεγάλα είναι τα κέρδη. Επομένω. Έτσι θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα. Είναι θέμα δικαιοσύνης. Είναι θέμα ηθικό τελικά. Όπως δεν μα αρέσει η κλοπή, επίσης θα πρέπει να μα δυσαρεστεί το ότι οι γυναίκες δεν αμείβονται όσο θα έπρεπε. Θα πρέπει να θεσπιστούν και κάποιε κυρώσεις. Τέλο το θέμα είναι διαστατικό. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή Σύντομα όμω για να μπορέσουμε να πάρουμε και άλλε ερωτήσει. Σα ευχαριστώ. Δεν Θα πρέπει να ξεχνούμε ότι έχουμε εδώ πέρα δύο διαστάσει. Είναι διτό το, το, το ζήτημα και αυτέ οι δύο διαστάσει ε, είναι αλληλένδετε και δεν θα πρέπει επομένω να γνώμω ούτε τη μία ούτε την άλλη. Πρώτα ε, την πτυχή τη ισότητα και των δικαιωμάτων ότι δηλαδή είναι θέμα ισότητα ευκαιριών, είναι θέμα ισότητα μεταξύ φυσικών προσώπων τελικά τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι δυνατόν όλα να, να, εξετάζονται από πλευρά οικονομική και οικονομίστικη. Δηλαδή, μπορεί κανεί να έχει δίκαιη δίκη, μπορεί να, αυτό να έχει αναγνωριστεί στην Ευρώπη σαν θεμελιώδη δικαίωμα, όμω κανένα δεν κάθεται να, να, να, πει πόσο κοστίζει, πόσο ωφελεί ε, το να έχουμε δίκαιη δίκη. Όμω, από την άλλη μεριά, βεβαίω και υπάρχει η πτυχή. Ε, οικονομική, επιχειρηματική, στο θέμα της ισότητας. Σας παραπέμπω στο δελτίο τύπου της Δευτέρας. Θα πάνε καλύτερα οι επιχειρήσει. Έχουν περισσότερη ανταγωνιστικότητα, περισσότερα κέρδη όποτε έχουμε ισότητα. Έχουμε την έκθεση McKinsey και κατελήξε στο ότι 56% μεγαλύτερα κέρδη έχουν οι εταιρείε όπου έχουν περισσότερη ισορροπία. Οι 290 εταιρείε εισηγμένε, η κοίταξη Έρνη Young και κατέληξε στο Διοικητικό Συμβούλιο, υπήρχε τουλάχιστον μία γυναίκα και όλε αυτέ οι εταιρείε τα πήγαν καλύτερα από εκείνε που δεν είχαν ούτε μία γυναίκα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σα ε, παραπέμπω επίση και σε, αυτή, σε αυτό το κείμενο τη ε, της, της, της Δευτέρα όπου εκεί πέρα υπάρχουν ένα σωρό παραπομπέ από ειδικέ πηγέ, εξειδικευμένε πηγέ για το θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρο, και δίνει το λόγο στον επόμενο που έχει ζητήσει. Γιάννα Σούλτ, ελεύθερη δημοσιογράφος από τη Γερμανία. Πρώτη ερώτηση που αφορά στατιστικά στοιχεία. Σε ποιες χώρες, σε ποια χώρα υπάρχει το μεγαλύτερο χάσμα και αυτό από τι μπορεί να οφείλεται. Δεύτερον, δεύτερη ερώτηση, η Επιτροπή δεν είναι σήμερα υποχρεωμένοι, δεν υπάρχουν δηλαδή νομοθεσίες στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προκαλούν αντιδράσεις, όπως παραδείγματος χάρη αυτές που είδαμε στη Γερμανία σε σχέση με τις προτάσεις της κυρίας Ρέντινγκ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ερωτήσεις σας. Η δεύτερη ερώτηση σίγουρα απευθύνεται κατευθείαν στην Επιτροπή. Η άλλη ενδεχομένως μπορεί να απαντηθεί από τα μέλη του πάνελ. Η Σύρη μας λέει εδώ ότι το μεγαλύτερο χάσμα βρίσκεται στην Εστονία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί βέβαια να σας δώσει κάποιο απόσπασμα από αυτά τα στατιστικά δεδομένα, αλλά σας παραπέμπω στους ε, ευρωβουλευτές για, για αυτή τη δουλειά. Πάντως, για να σας ε, απαντήσω σε σχέση με τη σχέση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ του μισθολογικού χάσματος και της οικονομικής ε, συγκυρίας, εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι αυτόματο, αυτονόητο το ότι οι χώρες που βρίσκονται σε χειρότερη οικονομική κατάσταση ε, επίσης έχουν ε, μεγαλύτερο μισθολογικό χάσμα. Αυτό εξαρτάται από τις διαφορές της αγοράς εργασίας, εξαρτάται από την παράδοση του δικαίου κάθε χώρα. Τα είπαμε εδώ προηγουμένως. Κάποιες χώρες μέλη καθορίζουν τη μισθολογική πολιτική επί τη βάση των διαπραγματεύσεων των εργαζομένων. Άλλες χώρες έχουν άλλου είδους ε, ενδελεχή κλίμακα μισθολογική, συντελεστές, ανάλογα με τη δουλειά του καθένα κλπ. Οπότε αυτό οδηγεί σε μικρότερο μισθολογικό χάσμα. Για να απαντήσω τώρα στην άλλη σας ερώτηση, λαγωνικά. Σας θυμίζω ότι τη Δευτέρα η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ δημοσίευσε μια έκθεση για το πώς έχει τώρα η κατάσταση στην Ευρώπη από πλευράς ε, ισορροπίας, η έλλειψη ισορροπίας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στα δικαιωτικά συμβούλια. Επίσης, έχει τονιστεί ότι η μέθοδος της θέσπισης ε, νόμων είναι μόνο μία από τις μεθόδους για να αρθεί αυτό το πρόβλημα. Και τέλος θα αποφασίζουν σχετικά οι επίτροποι με τα, την ολοκλήρωση της διαβούλευσης. Ευχαριστώ πολύ. Στο πρώτο σας ερώτημα, όσον αφορά τα αποτελέσματα των στατιστικών, η χώρα που έχει τις, μεγαλ... τις μικρότερες διαφορές σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat του 2009. Το έχει επεξεργαστεί η Μαρία Θά, μη προσαρμοσμένα στοιχεία. Είναι η Σλοβενία. Τη μεγαλύτερη, τη μεγαλύτερη διαφορά την παρατηρούμε στην Εστονία. Η Γερμανία είναι η τέταρτη ξεκινώντας από τα χειρότερα αποτελέσματα. Έχουμε την Τσεχία, την Αυστρία και κατόπιν τη Γερμανία. Αφού είστε Γερμανίδα, ε, φαντάζομαι σας ενδιαφέρουν τα στοιχεία που αφορούν τη χώρα σας. Ε, τα στοιχεία αυτά πρέπει να υπάρχουν στο φάκελό σας. Τα έχουμε δώσει γραπτά. Και βεβαίω συνεχίζουν να υπάρχουν σημαντικέ διαφορέ, σημαντικέ παραδόσεις από τη μία χώρα στην άλλη. Τα στερεότυπα υπάρχουν, αλλά δεν είναι τα ίδια παντού. Έχετε το λόγο. Εγώ είμαι δημοσιογράφος από το Αμβούργο. Θα ήθελα να μιλήσω για τις γυναίκες που έχουν ηγετικές ε, θέσεις. που βεβαίω μπορούν να ανταπεξέλθουν σε διάφορα επιπλέον έξοδα. Όλες οι γυναίκες όμως δεν έχουν αυτές τις ηγετικέ θέσεις, δεν έχουν υψηλούς μισθούς, άρα δεν μπορούν να ε, καλύψουν έξοδα που αφορούν τη φροντίδα των παιδιών, την εργασία στο σπίτι κτλ. Ναι, σας ευχαριστώ. Περβός. Μπορείς να απαντήσεις την ερώτηση αυτή. Γιατί νομίζω ότι αναφέρθηκε στο θέμα αυτό στην εισήγησή σου. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μίλησα για τις προτάσεις της κυρίας Ρέντινγκ λέγοντας βεβαίως ότι τα προβλήματα δεν πρόκειται να λυθούν ε, από τη μία μέρα στην άλλη. Η κυρία Κράτσα μίλησε όχι για το πράσινο ανατοτόριο, είπε όμως ότι πολλοί τομείς δεν καλύπτονται από τις γυναίκες. Όπως παραδείγματος χάρη, πολλές φορές αρκετές γυναίκες δεν είναι υποψήφιες για πολύ σημαντικές ηγετικές θέσεις, υψηλές θέσεις. Εγώ μπορώ να πω όμως και το αντίθετο, ότι υπάρχουν θέσεις για τις οποίες υπάρχουν πάρα πολλές υποψήφιες γυναίκες. Τι εννοώ τις χρηματαγορές με το που υπάρχει μία πρόταση παραδείγματος χάρη για να επιβληθεί ένας φόρος η απάντηση είναι αν κάνετε αυτό, αν επιβάλλετε αυτό το φόρο παραδείγματος χάρη όλα τα κεφάλαια θα φύγουν από την Ευρώπη παραδείγματος χάρη. Και το ίδιο επιχείρημα πολλές φορές βλέπουμε όταν δεν υπάρχει παραδείγματος χάρη μια υποψήφια γυναίκα, η απάντηση είναι «Α, μα δεν υπάρχουν υποψήφιες γυναίκες να καλύψουν τη θέση αυτή». Μα κοιτάξτε, υπάρχουν όμως και άλλες κατηγορίες και άλλες θέσεις όπου υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες. Κοιτάξτε τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι γραμματείες των επιτροπών, παραδείγματος χάρη. Κοιτάξτε. Η ισορροπία των φίλων Και συγκρίνεται το με τις διευθύνσεις, τις υψηλές θέσεις στη διοίκηση. Στο Προεδρείο υπάρχει κάποια ισορροπία. Μπορεί να βελτιωθεί βεβαίως η κατάσταση πολύ περισσότερο, αλλά δεν πρόκειται να διορθωθεί το φαινόμενο αυτό με φυσικό τρόπο, αν δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ε, θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω κάτι, ε, παρόλο που ε, καταρχάς θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είχα πει και στην αρχή, ότι ήδη προτείνουμε ένα πλαίσιο συμπληρωματικών πολιτικών μαζί με τα κουότα που θα διευκολύνουν τις γυναίκες να αξιοποιήσουν και τις ευκαιρίες που δίνουν τα κουότα Θέλω να σας πω ότι έρευνες που, που είχα την ευκαιρία να ανακαλύψω προωθώντας την σύνταξη της έκθεσής μου, λένε ότι οι, οι οικογενειακές υποχρεώσεις δεν είναι το πιο σημαντικό στο πλαίσιο, στο επίπεδο που οι γυναίκες επιδιώκουν υψηλές θέσεις ευθύνης. Ίσως γιατί βρίσκονται σε μια ηλικία που έχουν περάσει η, έχει περάσει η έννοια της, της φροντίδας των μικρών παιδιών πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι καριέρες είναι απαιτητικέ. Οπουδήποτε και αν γίνονται. Στην πολιτική, στον επαγγελματικό βίο, στον καλλιτεχνικό ε, ή στον οικονομικό ενώ στον χώρο των επιχειρήσεων, στον χώρο των καλλιτεχνικών, οπουδήποτε κανείς θέλει. Άνδρας ή γυναίκα να χτίσει μια καριέρα πρέπει να επενδύσει πολύ, να κάνει θυσίες από τον εαυτό του, να έχει στρατηγικό στόχο, να ξέρει να επενδύσει και ε, χρειάζεται η φιλοδοξία και η δέσμευση και των ίδιων των γυναικών. Ποτέ και πουθενά δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Στόχος μας είναι να, να δημιουργηθούν οι συνθήκες και ευκαιρίες όπου οι γυναίκες εισάξια με τους άνδρες ονειρεύονται, κάνουν σχέδια, επιδιώκουν, στοχεύουν και επιτυχάνουν. Ποτέ δεν πρόκειται να λυθούν όλα τα προβλήματα και να γίνουν δρόμοι εύκολοι και στρωμένοι με δάφνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω άλλη ερώτηση. Και αυτό είναι μάλλον ευχάριστο, διότι φτάσαμε στο τέλος της πρωινής μας συζήτησης. Α, βλέπω μία ερώτηση. Κοιτάξτε, πρέπει η ερώτηση να είναι συγκεκριμένη σε ένα άτομο, αλλιώ στην Επιτροπή. Εντάξει, πολύ σύντομα παρακαλώ. Πατήστε και το κουμπί του μικροφόνου. Μιλάρα ναι, με λένε, είμαι Ισπανίδα δημοσιογράφος. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Ε, υποθέτω ότι το θέμα της ποσόστοσης ε, το έχουμε ολοκληρώσει. Ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ξέρετε ποιες χώρες ε, περίπου είναι κατά των ποσοστώσεων. Και δεύτερο, δεύτερη ερώτηση. Ε, προτίθεστε να, να οργανώσετε εκστρατείες με βασικούς αποδέκτες άντρες. Απάντηση. Ίσως είναι προώρο να αρχίσουμε να κατονομάζουμε κράτη-μέλη που είναι κατά και άλλα που είναι υπέρ ε, των ποσοστώσεων. Το Φεβρουάριο στο πιο πρόσφατο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων έγινε μια δημόσια ε, συζήτηση που αναμεταδόθηκε δηλαδή στο διαδίκτυο και πήραν εδώ λόγο εκπρόσωποι όλων των κρατών σχετικά με την ποσοστώσεις στα διοικητικά συμβούλια. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο, διότι έχει αρχίσει να γίνεται δημοφιλές το ζήτημα και θα έπρεπε να εξηγήσουμε διεξοδικότερα ε, το εξή ότι ε, δεν θεωρείται ότι όλα γίνονται για επικοινωνιακούς λόγους αλλά ε, αρχίζει να υπάρχει συνειδητοποίηση ότι πρόκειται για ένα στοιχείο μιας ευρύτερης πολιτικής ατζέντα και ξέρετε σε επίπεδο λήψης αποφάσεων υπάρχει εντατικός διάλογος όχι μόνο για αυτό το ζήτημα αλλά και για άλλα όπως η παρουσία των γυναικών όχι μόνο στα διοικητικά συμβούλια αλλά και σε διοικητικού χαρακτήρα θέσεις, δηλαδή ως στελέχη σχετικά υψηλόβαθμα των επιχειρήσεων. Επίσης, ε, ε, σχετικά με τις ε, εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, σα είπα ότι έχουμε την εκστρατεία. Τι γίνεται όμως οι υπόλοιπε εταιρείε ε, πέρα από τα χρηματιστήρια του Λονδίνου, της ε, του Παρισιού. Τι γίνεται στις υπόλοιπε επιχειρήσεις. Επίσης, η συγκεκριμένα η σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα. Ποια είναι η κατάσταση εκεί, ποιε είναι οι διαφορέ ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ποιε πολιτικές και ποιε προσαρμογές χρειάζονται οι εργοδότες ούτω ώστε στο εσωτερικό των επιχειρήσεών τους να μπορέσουν να επανισορροπήσουν την κατάσταση, να ε, ε, ανακτηθεί δηλαδή, ε, να επιτευχθεί μάλλον ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα σε επίπεδο επιχειρήσεων. Θα ήθελα εντάχει να απαντήσω και στο ερώτημά σα σχετικά με μια εκστρατεία με αποδέκτες βασικά του άντρε. Το έχουμε σκεφτεί και φυσικά τα δύο χρόνια έχουμε ήδη ξεκινήσει σχετικές προπαρασκευαστικές εργασίες. Έχουμε ήδη ζητήσει μελέτη που αναλύει σε επίπεδο βάσης κυρίως ε, στο εσωτερικό ε, δημοσίων και ιδιωτικών ε, επιχειρήσεων αναλύει το ρόλο των ανδρών για την επίτευξη του στόχου της μεγαλύτερης ισότητας ε, των δύο φύλων σε επίπεδο έργο, εργαζομένων σε αυτές τις δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες. Του χρόνου πιστεύω, αν θυμάμαι καλά, είναι που θα δημοσιοποιηθεί το πόρισμα αυτής της μελέτης. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Ε, καλή όρεξη θα ήθελα να σας ευχηθώ και θα επανέλθουμε στις 2 και 4. Σας ευχαριστώ όλους. Τα λέμε ξανά στις 2 και 4.